Η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί και θα περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Βάσει της ημερήσιας διάταξης θα ψηφιστούν ε, οι θανατικές ε, καταδίκες κατά του Δημήτρη Καναβαλιόφ και του κυρίου Καβαλιόφ. Έχουμε έξι ψηφίσματα, προτάσεις ψηφισμάτων θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές. Ε, γίνεται ομόφωνα δεκτό το ψήφισμα. Τώρα θα έρθουμε στο ψήφισμα για την Αίγυπτο. Έχουμε 7 ψηφίσματα και ένα κοινό ψήφισμα 7 πολιτικών ομάδων και εδώ δεν έχουν ε, κατατεθεί ε, τροπολογίες. Ποιος είναι υπέρ του ψηφίσματος. Κατά αποχές και, αυτή, αυτό το ψήφισμα εγκρίνεται ομόφωνα. Βάσει τη σημερινή διάταξη, τώρα έχουμε τη ψηφοφορία για έξι ε, ψηφίσματα για την θανατική ποινή στην Ιαπωνία και έχουμε και ένα κοινό ψήφισμα. Ο κύριος Τσίσεστερ επί διαδικαστικού. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ε, ε μπερδεύτηκα κάπως γιατί υπήρχε ένα, με πρόταση ψήφισματο από την Ευρώπη τη Ελευθερία και Δημοκρατίας ε, πριν από το κοινό ψήφισμα. Ε, μπορείτε να μου το διευκρινίσετε αυτό το σημείο, γιατί εγώ ψήφισα σύμφωνα με αυτό που νόμιζα. Κύριε Τσίριστερ, είχαμε ένα ψήφισμα του ΕΦΤΕ για την Ιαπωνία, αλλά είμαστε ακόμα στην Αίγυπτο, δεν έχουμε φτάσει στην Ιαπωνία έχουμε έξι ψηφίσματα και ένα κοινό ψήφισμα πέντε πολιτικών ομάδων. Τώρα θα ψηφίσουμε λοιπόν, ε, προηγουμένως θα ψηφίσουμε το κείμενο του EFD. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα θα έρθουμε στο κοινό ψήφισμα πέντε πολιτικών ομάδων. Δεν έχουν κατατεθεί τροπολογίες. Άρα λοιπόν θα ψηφίσουμε για το σύνολο του κειμένου με οριστική ψηφοφορία. Με ονομαστική ψηφοφορία, συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε άπαντε. Πέρα της ψηφοφορίας. Το ψήφισμα έγινε δεκτό. 43 ε, ψήφοι υπέρ. Ε, τέσσερις αποχές, κατά τα άλλα είναι ομόφωνο το αποτέλεσμα. Τα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης θα υποβληθούν στην προσεχή συνεδρίαση προς έγκριση. Δεν υπάρχουν καθόλου ενστάσεις για αυτά τα ψηφίσματα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Κυρία Κορόλα, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ήθελα απλώς να πω ότι ψήφισα υπέρ, αλλά η κονσόλα δεν λειτουργούσε. Θα συμπεριληφθείτε στα πρακτικά, κυρία Κορόλα. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους καλή επιστροφή στα σπίτια τους. Στην περίπτωση που ε, λόγω δυσχερών κλιματικών συνθήκων η απεργία στη Γερμανία ε,